Okay, uh, welcome back uh, Χαίρετε. Καλώς ορίσατε και πάλι στη συνεδρία της Επιτροπής. Θα ξεκινήσουμε τώρα. Θα ξεκινήσω σου λοιπόν. Λοιπόν, σας καλωσορίζω να περάσουμε στο σημείο 11 της σημερινής διάταξης. Ε, είναι στην ουσία το σημείο 10 αφορά τις ε, συνθήκες απασχόλησης ε, των υπαλλήλων και άλλων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αλλαγές που γίνονται στο, στο καταστατικό δημοσιοπαλληλικής καταστάσεως. Ευχαριστώ, λέει κυρία Κοχμέριν. Ναι, μεν ε, φαίνεται τεχνικό το θέμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είναι η μεταρρύθμιση του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως που αφορούν περίπου που αφορά ο κανονισμός 55.000 περίπου υπαλλήλους δεν αφορά μόνο την ε, το προσωπικό που έχουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αφορά και όλα τα θεσμικά όργανα. Κοινοβούλιο, Επιτροπή Συμβούλιο, Επιτροπή Περιφερειών, Δικαστήριο, περίπου 55.000. Καθορίζει τους κανόνες για τους όρους εργασίας, ε, τη συνταξιοδότηση, όλα τα θέματα που αφορούν την ε, ζωή εργασία των υπαλλήλων, την ε, εργασία των υπαλλήλων, την εργασιακή ζωή. Βέβαια είναι ιδιαίτερα ογκώδες εμείς το εξετάζουμε μόνο από πλευράς της ε, Επιτροπής Γυναικών. Γιατί γίνεται αυτή η μεταρρύθμιση, γιατί υπάρχουν κάποιες δημοσιονομικές ανησυχίες από πλευράς κρατών μελών, θέλουν να μειωθεί ο προϋπολογισμός των ε, Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων για το προσωπικό τους, θέλουν να μειωθεί η δαπάνη μέχρι το 2020 κατά 8 δις, σημαντικό ποσό, θέλουν να εφαρμοστεί ή τουλάχιστον να αποφασιστεί η μεταρρύθμιση φέτος, γιατί αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή που αποφασίστηκε το 2004 θα εξακολουθήσει να ισχύει, κάτι που θα αυξήσει κατά 5% τον προπολογισμό για τις δαπάνε αυτές. Το αντίθετο από αυτό που επιδιώκουν. Πιέζει ο χρόνο λοιπόν, το Κοινοβούλιο έχει προετοιμαστεί πολύ καλά, εργαστήκαμε ταχύτατα για το θέμα αυτό όταν υποβλήθηκε η πρόταση από τον αντιπρόεδρο Σεύτοβιτ για πλευρά, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εξέτασαν διάφορε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Οι κύριε προτάσει για περικοπέ από πλευρά τη Κομισιόν ήταν, α πούμε, ένα κούρεμα κατά 5% του προσωπικού και άλλα στοιχεία αύξηση των ωρών εργασίας εβδομαδιαίως αύξηση της ηλικία της ταξιοδότησης και δημιουργία μιας νέας κατηγορίας χαμηλοαμοιβόμενων εργαζομένων, χαμηλόμισθων. Επί της ουσίας αρμόδια είναι η Νομική Επιτροπή. Η Επιτροπή Προπολογισμών και Ελέγχου έκανε γνωμοδότηση, όπως και εμείς. Η Επιτροπή Απασχόλησης έστειλε μία επιστολή και η κυρία Περές Έστειλε λοιπόν αυτή την επιστολή με την οποία ε, συμφωνώ θα μπορούσαμε να την υποστηρίξουμε κι εμείς. Είναι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που ασχολείται με το θέμα αυτό, δηλαδή Υπουργοί Εξωτερικών. Είναι σαφές ότι έχουν δημοσιονομικές προτεραιότητες. Τα σημεία κλειδιά για μας είναι να βρούμε τρόπο για να γίνουν αυτές οι εξοικονομήσεις τα στοιχεία που προτείνονται πρέπει να εξεταστούν από την Επιτροπή μας σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στην πολιτική για ισότητα των φύλων. Γενικά μπορούμε να υποστηρίξουμε τις περισσότερες προτάσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ένα περιβάλλον εργασίας σύγχρονο και αποτελεσματικό από πλευράς κόστους και εφόσον στα κράτη-μέλη ζητάμε να εργάζονται περισσότερο, για παράδειγμα από τα 63 στα 65 με δυνατότητα να μείνουν μέχρι τα 67 υπάλληλοι των θεσμικών οργάνων δεν είναι υπερβολικό. Δεν είναι υπερβολική απέτηση έναντι του προσωπικού. Ποια θέματα λοιπόν έχει η Επιτροπή μας. Κυρίως εξέτασα τα ζητήματα που αφορούν την αρχή ισότητα των φύλων και το συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματική ζωής. Αυτά είναι δική μας αρμοδιότητα. Με χαρά στην επιστολή της κυρίας Μπερέζ βλέπω ότι και εκείνη αναφέρει μερικά σημεία που σχετίζονται με αυτό. Αν και βέβαια για κάποια μπορούμε να έχουμε κάποιες επικρίσεις. Πρώτον, χρειαζόμαστε σύγχρονες συνθήκες εργασίας για υψηλά ειδικευμένο προσωπικό, όπως το χρειαζόμαστε. Και όταν λέμε σύγχρονε συνθήκε εργασία, ένα σημαντικό στοιχείο είναι να υπάρξει το πλαίσιο για το συνδυασμό προσωπική και οικογενειακή ζωή και για τα δύο φύλλα. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι τα περισσότερα μέτρα που εφαρμόζονται τα αξιοποιούν οι γυναίκε. Όχι μόνο επειδή τα δύο φύλλα έχουν διαφορέ προτεραιοτήτων, αλλά γιατί έχει επιπτώσει στα διαδρομία. Πρέπει λοιπόν αυτό να το, μετατρε... να το μεταρρυθμίσουμε. Αυτό αφορά τη μερική εργασία, την τηλεεργασία, το ελαστικό ωράριο. Εδώ πρέπει να γίνουν βελτιώσεις και στην ε, γνωμοδότησή μου που έχετε στο φάκελό σας βλέπετε τις προτάσεις μου. Το άλλο σημείο είναι η γονική άδεια. Τι σημαίνει για να το πω απλά. Είναι τέτοιες οι προϋποθέσεις που αποθαρρύνει τις αιτήσει. Η διάρκεια είναι έξι μήνες. Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Αν κάποιος έχει ε, διάθεση να υπάρξει τροπολόγηση για το θέμα αυτό, παρακαλώ. Εγώ κοιτάζω περισσότερο την οικονομική πλευρά της γονικής άδειας. Μέχρι τώρα το ποσό προσαρμόζεται με βάση 780 ευρώ. Οπότε στην ουσία καταλήγουμε σε περίπου 900 ευρώ. Αν δείτε την πυραμίδα αμοιβών στην Ένωση, είναι απαγορευτικό. Δεν είναι δυνατόν να πάρει κανείς γονική άδεια και να ζήσει με 900 ευρώ. Αν έχει οικογένεια, αν είστε ε, η κύρια πηγή εισοδήματος της οικογένειας. Στα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν πολλές ανησυχίες ε, για τις δαπάνες του προσωπικού, στα κράτη-μέλη γίνεται διαφορετικά. Πληρώνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό του μισθού σας έως κάποιο ανώτατο όριο. Αυτό θα πρότεινα και εγώ για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Θα πρότεινα ε, ένα μικρότερο ποσοστό από τα ποσοστά που βλέπουμε στα κράτη-μέλη που είναι 60% και έναν τρόπο υπολογισμού με βάση τα διάφορα στοιχεία του βαθμού των υπαλλήλων. Κυρίως ε, τους βαθμούς ε, που κυρίως έχουν ε, τα άτομα που κάνουν παιδιά. Και φτάνουν σε ένα ποσό 2.500 ευρώ. Είναι ουσιαστική διαφορά. Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις ωστόσο δεν είναι τόσο σημαντικές. Διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για 6 μήνες, η περίοδος είναι μόνο εξαμηνιαία Έγιναν υπολογισμός και θεωρήσαμε ότι η επίπτωση θα είναι περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ. Αν το συγκρίνουμε με την πολιτική σημασία μιας σωστής γονικής άδειας, δεν είναι τόσο μεγάλος αριθμός. Συνέχεια λέμε στην κοινή γνώμη ότι η γονική άδεια πρέπει να είναι κάτι που να μπορούν να το πάρουν και άνδρες και γυναίκες για ισότητα των φίλων, να μην δημιουργεί πρόβλημα στα υδρομή των γυναικών εκ των υστέρων κτλ. Αυτή τη στιγμή μόνο 8% παίρνει γονική άδεια. 80% από αυτούς είναι γυναίκες ε, χαμηλόμιστες. Ένα άλλο στοιχείο δεν συμπεριλαμβάνεται ακόμη στο σχέδιο γνωμοδότησης, αλλά νομίζω ότι αντιμετωπίζεται σε άλλες τροπολογίες, είναι αυτή η νέα ομάδα χαμηλομίστων, που καταργήθηκε πριν από μερικά χρόνια, διότι διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα άτομα που εργάζονταν εκεί είχαν προσόντα όπως και οι πιο υψηλόμιστοι. Απλώς αντιμετωπίζονταν με άλλον τρόπο. Και ήταν κυρίως γυναίκες. Όταν μιλάμε λοιπόν για το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, δημιουργούμε τώρα εμείς ένα τέτοιο χάσμα εδώ, στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να το σχολιάσουμε αυτό και να το επικρίνουμε έντονα. Μερικά μικρότερα θέματα. Δεν θα πρέπει μόνο να στέλνει ένα εσωτερικό σημείωμα ο Γενικός Γραμματέας για να υπάρξει δυνατότητα σωστού θυλασμού. Και επίσης να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της εγκυμοσύνης. διότι με, βάση τον κανονισμό είναι δυνατόν να απολύσεις μία έγκυο γυναίκα. Δεν μπορείς να την απολύσεις μόνο αν είναι σε άδεια τοκετού και μητρότητας. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε κάτι τέτοιο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Να περιοριστώ σε αυτά, προσβλέπω στα σχόλιά σας και φυσικά να απαντήσω αν μπορώ τις ερωτήσεις σας. Καταληκτικά ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μην θεωρείται ότι μόνο επιβάλλουν υποχρεώσεις και κάνουν συστάσεις στους άλλους για θέματα ισότητας των φύλων και το συνδυασμό καριέρας και οικογενειακής ζωής, πρέπει και να εφαρμόζουμε αυτά τα οποία κηρύττουμε. Να παίξουμε το ρόλο προτύπου. Αν θέλουμε να κάνουμε, όπως είπε και ο Γκάντι, τις αλλαγές που θέλουμε στον κόσμο πρώτα στον εαυτό μας. Να μην θεωρήσουμε λοιπόν ότι δεν είναι αρκετά σημαντικό αυτό το θέμα και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε έχετε το λόγο παρακαλώ να υπογραμμίσω ότι δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Στις 5 έχουμε την κοινή μας συνεδρίαση όπου θα ψηφίσουμε. Έχουμε πάρα πολλέ ε, τροπολογίε να ψηφίσουμε. Πρέπει να τελειώσουμε πριν τι 5 γιατί έχουμε και άλλο ένα θέμα να συζητήσουμε. Παρακαλώ, το έχετε υπόψη σας όταν πάρετε το λόγο. και μετά Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που ήρθε στη συνεδρία των τονιστών η Σιβάνα και ήδη συζητήσαμε το θέμα αυτό. Πολύ σημαντικό η Επιτροπή Γυναικών να συντάξει γνωμοδότηση διότι δουλεύουν πολλές γυναίκες στα θεσμικά όργανα της Ένωσης ε, αν δούμε βέβαια και τις σχέσεις ισχύω, δεν τα πάμε τόσο καλά. Υπάρχουν πολύ λιγότερες γυναίκες στις ηγετικές θέσεις. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ την εισηγήτρια για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και υπογραμμίζω τρία πολύ σημαντικά. το νέο βαθμό ASTSC στην αρχική πρόταση είναι πολύ χαμηλόμιστη και θα θίξει κυρίως τις γυναίκες. Δεν με ικανοποιεί όπως έχει τώρα η κατάσταση. Γιατί οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε αυτό το βαθμό θα είναι γυναίκες. Δεν καταλαβαίνω τι βαθμούς έχουν δημιουργήσει. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το κρατήσουμε ή να υπάρξει κάπως πιο υψηλόμιστη, να υπάρξουν κάπως πιο υψηλόμιστοι ε, βαθμοί. Το ελαστικό ωράριο για όλους. Βεβαίω, η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο είναι υπέρ της ισότητας. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά έναν βοηθό από έναν ευρωβουλευτή. Να υπενθυμίσω ότι αυτά που κάνουμε αποτελούν υπόδειγμα για τους άλλους. Καταλαβαίνω, υπάρχει κρίση. Και ότι θα πρέπει να μειωθούν κατά 5% οι πάλι στο μέλλον. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να είμαστε και λογικοί, να κρατήσουμε υπαλλήλου ποιότητας. Και βεβαίω ξέροντας ότι 60% των γυναικών πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο παίζει ρόλο. Για τη γονική άδεια συμφωνώ με την αντιμετώπιση σας. Από μια συζήτηση που κάναμε με την Dagmar Rod Merem, την κυρίω εισηγήτρια, καταλάβαμε ότι θα υποστηρίξει μόνο την τροπολογία για την ισότητα φίλων και το συνδυασμό οικογένειας και σταδιοδρομία στη φροντίδα για τα παιδιά και την τροπολογία 4 για την ε, ισότητα φύλων. Στην έκθεσή της κάνει μια τροπολογία για ένα νέο βαθμό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα, αλλά φυσικά θα πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι τέλους για αυτό το θέμα. Αλλά ε, τι ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Συζητήσαμε την ε, δυνατότητα να υποβάλουμε τροπολογία για να απαγορεύεται να απολύονται εργαζόμενες κατά τη διάρκεια της ε, εγκυμοσύνης. Για την τελεργασία η Ντάγμαρ είναι κατά, γιατί λέει ότι θα είναι πολύ δύσκολο να μπει στον κανονισμό, ότι θα επιστρέψουν οι γυναίκες στο σπίτι και θα αυξηθεί η ανισότητα. Μα δεν μιλάμε μόνο για γυναίκες, αλλά και για άνδρες. Δεν νομίζω ότι μόνο οι γυναίκες θα έπρεπε να εποφελούνται από την τηλεργασία. Το να εργάζεται κανείς από το σπίτι δεν σημαίνει ότι απλώς κάνεις τον οικοκυριό Και έδωσε τις εξής εξηγήσει. Βεβαίως πρέπει να υπάρξουν εξοικονομήσεις, αλλά δεν είναι σωστή η προτεραιότητα αυτή. Το θέμα είναι να υπάρχει σωστή αντιμετώπιση και να βρούμε τα χρήματα για αυτή τη σωστή αντιμετώπιση. Αν είδατε και τα κείμενα που μας έστειλαν τα συνδικάτα σε διάφορους, τίθεται και άλλα θέματα. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των ε, συντάξεων, που θα τις μειώσει κατά 30% σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους. Και αυτό θα θίξει πολύ περισσότερες γυναίκες παρά τους άνδρες. Και επειδή υπάρχει ήδη χάσμα συντάξεων όπως αναφέρθηκε, πρέπει να υπογραμμίσουμε αυτό το πρόβλημα η κυρία συγγήτρια είπε ότι δεν θα την υποστηρίξει, αλλά επειδή εμείς ασχολούμαστε με αυτό το χάσμα μισθών, αμοιβών, είναι, τίθεται θέμα και χάσματος συντάξεων. Άρα πρέπει να εμείνουμε. Αλλά αυτή είναι η γνώμη της συζητήτριας, εάν θα θέλατε να συζητήσετε μαζί της. Ευχαριστώ. σε περίπου 7 λεπτά θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης. Οπότε άλλοι δύο σύντομα μπορούν να μιλήσουν, Κορνέλισεν και Λούλινγκ. Κορνέλισεν παρακαλώ πρώτα. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Όπως είπα και στις συνεδρίες των συντονιστών, ε, την έκθεση αυτή την ε, αντιλήφθηκα λίγο καθυστερημένα. Θα ήθελα περισσότερο χρόνο για να τη μελετήσω. Είναι πολύ πλούσιο το υλικό που πρέπει να σκεφτεί κανείς. Αλλά επειδή πρόκειται για γνωμοδότηση, εάν μας έρθει κάποια εξαιρετική ιδέα, μπορούμε να τις υποβάλουμε σε μορφές τροπολογιών από κοινού με μέλη της Γιούρη, δηλαδή προς την Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή. Ας το έχουμε και αυτό κατά νου. Μερικές σύντομες παρατηρήσεις. Κάποια πράγματα θα πρέπει να διορθωθούν, όπως να υπάρχει χώρος για τον αθυλασμό, ε, για το μετρικό γάλα, Αυτά θα μπορούσαν να υπάρχουν και στην κυρία οδηγία ή και σημαντικότερα ζητήματα οπω στόχη για τι γυναίκε στα υψηλότερα κλιμάκια, στόχος για την κάλυψη του χάσματος ε, των αμοιβών ε, για του υπαλλήλου. Δηλαδή αυτά που συνήθως συνιστούμε στον έξω κόσμο να φροντίσουμε να ισχύουν και για τον δικό μας. Ε, για την χαμηλόμεστη ομάδα είπατε να φανούμε επικριτικοί εδώ. Δηλαδή να διαφωνήσουμε πλήρως, να ζητήσουμε να μην υπάρχει αυτή η ομάδα ή έχετε κάποιες αναλλακτικέ προτάσεις. Και για την μερική εργασία. Ε, για τους λόγους που επιτρέπουν να ζητήσει κανείς κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε, πιστεύω, να μην χρειάζεται τέτοια διολόγηση για τη μερική εργασία. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς να το ζητάει χωρίς ιδιαίτερη αιτιολόγηση. Ευχαριστούμε κυρία Λούλιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα πρέπει να σας ε, εκφράσω την έκπληξή μου που έμαθα ότι ε, ο εισηγητής έρχεται να δει τους συντονιστές πριν δει τους σκιώδει εισηγητές. Υπάρχει μια νέα διαδικασία σε αυτή την ε, Επιτροπή. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την ομάδα μου. Θα προτιμούσα λοιπόν να είχα ειδοποιηθεί ώστε να λάβω τα απαραίτητα μέτρα. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, διότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να σας πω απλούστατα κατά πόσον συμφωνώ. Τροπολογία 1. Θα μπορούσα να συμφωνήσω, διότι υπάρχουν περισσότερες γυναίκες από ότι άντρες αυτή τη στιγμή. Να το θυμόμαστε από την άποψη των επαλλήλων του Ευρωκοινοβουλίου. Θα χρειαστεί λοιπόν μάλλον θετική δράση και για του άντρε. εφόσον το επιτρέψουμε αυτό. Για την τροπολογία 2 και 3 όχι και όχι, 4 ναι, 5 όχι, 6 και 7 όχι. Δεν θα εξηγήσω τώρα την καθεμιά ξεχωριστά. Θα το κάνω εν ευθέτω χρόνο. Σίγουρα θα μας δοθεί ευκαιρία. 8 δεν είναι πραγματικό μέτρο συμφιλίωσης, διότι διοδρομία και το θυλασμός είναι ανά δύο εννέα να είμαστε προσεκτικοί, δέκα ε, όχι, έντεκα είναι διχασμένες εδώ οι απόψεις. Μήπως μάλιστα χειροτερέψουμε τα πράγματα για τους γονείς από ό,τι τώρα, σε σχέση με την άδεια του κετού. 15 είναι πολύ αμφίσιμη η τροπολογία. Κύριε Πρόεδρε, λίγο πολύ, επειδή δεν έχουμε και χρόνο, αυτή ήταν ε, η τοποθέτησή μας. Δεν έχω χρόνο να εξηγήσω την άποψή μας ε, λεπτομεριακά, αλλά θα το κάνω σε άλλη φάση, όταν ελπίζω ότι θα έχουμε μια πιο εντελεχή συζήτηση. Ευχαριστώ. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο πλέον. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Εάν δεν είχαμε την κοινή ψηφοφορία με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, θα το συζητούσαμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Όντω, είναι κρίμα που δεν έχετε χρόνο να εκφραστείτε. σω κάτι να έχει να πει ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώ, πολύ σύντομα να πω ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί συνέχεια τη μεταρρύθμιση του 2004 που επέτρεψε να γίνουν βήματα προόδου στον τομέα των ίσων ευκαιριών και της προστασίας των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονίμων υπαλλήλων. Να θυμίσω ότι η τωρινή πρόταση θέλει να ανανεώσει την μεθοδολογία υπολογισμού προσαρμογής των μισθών και το τι γίνεται με τις ειδικέ ε, εισφορές. Στην ε, πρόταση αυτή έχουμε προβλέψει την έννοια του ελαστικού ωραρίου, κάτι που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο καταστατικό των υπαλλήλων. Γι' αυτό και κάποιες τροπολογίες από όσες έχουν επιβληθεί ε, αφορούν πρακτικέ που ήδη ισχύουν σε κάποια θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια για αυτό που τονίζει ότι κάποια μέτρα πραγματικά ήδη εφαρμόζονται από τα θεσμικά όργανα. Κατά τα άλλα, για τι τροπολογίε που θα έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις, θα φροντίσουμε να τις αναλύσουμε στο πλαίσιο του συνολικού πακέτου για τι εξοικονομήσει για το υπολογισμό του αντικτύπου των μέτρων. Κάτι που και η ίδια συγκέντρια το υπογράμμισε. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Eh, Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Κοχμερή για να κλείσω. Ευχαριστώ. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομη. Να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους συναδέλφους που ε, αφιέρωσαν τον χρόνο τους και διάβασαν την έκθεση και για το ε, πνεύμα συνεργασίας που δείχνουν. Όντω υπάρχουν κάποιε πτυχέ που μπορεί όντω να μην τύχουν ε, τη πλειοψηφία τη Επιτροπή ε, Νομικών Υποθέσεων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρουν την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, στο σύνολό του. Οπότε α μην αποθαρρυνόμαστε από τι ψηφοφορίε στην Επιτροπή Γιούρη. Ξέρω, α πούμε, ότι ο εισηγητή από την Επιτροπή Προπολογισμών έχει πολύ θετική άποψη για τι προτάσει, για τι αλλαγέ, για τη γονική άδεια. Και η Επιτροπή Προπολογισμών ε, προφανώ είναι και αυτή που θα πρέπει να μελετήσει τα αριθμητικά στοιχεία. Επίσης δεν άκουσα ένα απόλυτο όχι από την Κομισιόν, οπότε ας είμαστε κι εμείς σταθεροί στις δικές μας ε, απόψεις και ας υπερασπιστούμε αυτό που πιστεύουμε. Τώρα, σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν, συντάξεις ας πούμε, ή η χαμηλόμισθη υπάλληλη, η ομάδα των χαμηλόμισθων, έχουμε την προθεσμία πέμπτη μεσημέρι για την ομάδα των χαμηλόμισθων θα πρότεινα να κυκλοφορήσει η τροπολογία ανάμεσα στους ε, σκιώδες, να, δείτε, να τη δείτε, να πείτε τι, ποια είναι η άποψή σας. Η κυρία Ροτμπέρεντ έχει αλλάξει λιγάκι την ε, πρόταση κομισιόν, αλλά μπορούμε να την ξαναδούμε και εμείς. Και πάλι ευχαριστώ πολύ τους ε, συναδέλφους και ευχαριστώ που αφιερώσατε το χρόνο σας για την έκθεση αυτή. Και εγώ ευχαριστώ. Να σας πω λοιπόν ότι η προθεσμία για την αποβολή τροπολογιών στο κείμενο λέει 29 Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Η γραμματεία μας έδωσε την ευλογία της και μπορούμε να το επεκτείνουμε λίγο. Οπότε 29 Μαρτίου μέχρι τις 5 το απόγευμα η προθεσμία σας για την υποβολή των τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε στις 24 Απριλίου στην Επιτροπή. Η Γιούρη θα ψηφίσει την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω πότε θα πάει ακριβώς στην Ολομέλεια. κλείνουμε λοιπόν το σημείο 8. Πάμε στο σημείο 12. Μικρής κλίμακας και παραδοσιακή αλληλεία και η μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Η κυρία Ματέρα θα έπρεπε να είναι εδώ, να πάρει το λόγο. Λείπει όμως, δυστυχώς, δεν μπορεί να είναι παρούσα. Οπότε η κυρία Μπάουερ είναι αυτή που θα πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you so much on behalf of... Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη συναδέλφου να σα παρουσιάσω την γνωμοδότηση. Η συμβολή των γυναικών στην αλληλεία και στην υδατοκαλλιέργεια στο σχετικό τομέα είναι σημαντική. Ο ρόλο του ακόμη δεν έχει αναγνωριστεί όπω πρέπει. Όπως ε, είπε η Επίτροπος ε, Αλληλείας Μαρία Δαμανάκη, 31% ε, των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας τη της είναι γυναίκες. 56% αυτών εμπλέκονται και σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητε αλληλευτικές και οι γυναίκες επίσης δουλεύουν πάνω στα σκάφη σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας παραγωγής, από την αλίευση των ψαριών μέχρι την συλλογή των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, την αποστήρωση, επίσης πολλές είναι ιδιοκτήτριες καφών και λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, ο τομέας της αλίας θεωρείται αποκλειστικά τομέας που είναι καλός για σκληροτράχυλους ε, ναυτικούς, και οι γυναίκες ε, δυστυχώς την χάνουν διακριτικής μεταχείρισης όταν, ε, έχουν, ε, όταν παρεμβαίνουν. Το επαγγελματικό τους καθεστώς βεβαίως δεν αναγνωρίζεται, δεν έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά ωφέλη που πρέπει να τους παρέχει η ευθέση εργασία τους, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα Είναι πραγματικά σοκαριστικό που βλέπουμε ότι σε πολλούς λιμένες κάποια ελευτικά σκάφη δεν έχουν γυναική αποδητήρια. Στο ιστορικό της Ένωσης, γυναίκες από την Κύπρο, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ολλανδία ακόμα είναι οι μοναδικές που δεν έχουν καμία νομική αναγνώριση ε, του καθεστώτος τους. Κάποιοι έχουν, κάποιες έχουν θεωρηθεί ως ε, συνεργάτες της οικογενειακής επιχείρησης. Στη Γαλλία ε, ειδικό καθεστώς αλίας έχει δημιουργηθεί πια. Άλλες τώρα χώρες έχουν αναγνωρίσει το καθεστώς των ε, αυτοπασχολούμενων εργαζομένων γυναικών. Αυτό είναι κατάστη εφικτό λόγω της εφαρμογής της οδηγίας του 86 και της μεταγενέστερης οδηγίας 41 του 2010 όπου υπάρχει η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ, των, ε, ε, μεταξύ των και γυναικών στις δραστηριότητες αυτές. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των κρατών μελών υπάρχουν ασυνέπειες στις πολιτικές τους. Αυτές οι διαφορές ε, προκύπτουν, ε, φαίνονται μάλλον και ανάμεσα στην, ε, στις διάφορες περιφέρειες της ίδιας χώρας. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από τη Γαλλική ας πούμε, από τη Γαλλική νομοθεσία προκύπτουν τέτοιες ασυμβατότητες όπου υπήρξε η εισαγωγή μιας, ενός πιστοποιητικού συνεργαζόμενων των, των, των συζύγων των ναυτικών ως συνεργαζόμενων. Μία από τις προτεραιότητες της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών είναι να εγγυηθούν την κοινωνική και νομική προστασία των γυναικών που δουλεύουν σε τέτοια παραδοσιακή και μικρής κλίμακα αλληλεία, ώστε αυτό να διευκολύνει την συνέπεια μεταξύ των μισθών και άλλων των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, προστασία στην εργασία, κοινωνική προστασία. Βεβαίως πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα, για παράδειγμα η ενθάρρυνση και η ενίσχυση των ε, διαφόρων ενώσεων που παίζουν ρόλο σε αυτόν τον τομέα, καθώς επίσης και η παροχή οικονομικών κινήτρων για την, από το Ταμείο Αλίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρωμέβα έχει το λόγο. Just to be very brief. Θα είμαι πολύ σύντομος. Χαιρετίζω την εργασία που έκανε η συνάδελφός μας Ματέρα, που παρουσίασε η συνάδελφος Μπάουερ Τρεις τροπολογίες θα μπορούσα να προτείνω. Να κάνουμε συγκεκριμένη αναφορά στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. όπου να συμπεριλάβουμε την αρχή της ισότητας ευκαιριών. Να την υπογραμμίσουμε. Δεύτερον, Κάτι που επανειλημμένα έχουμε τονίσει, αλλά πρέπει να επιμείνουμε, πιστεύω. Να ζητήσουμε ε, χωριστές στατιστικές αναφύλω. Να ξέρουμε δηλαδή σαφώς τα διάφορα επίπεδα απασχόλησης και υποαπασχόλησης. Αναφύλω. Και τρίτον, η συμμετοχή των γυναικείων οργανώσεων στις ε, λεγόμενες συμβουλευτικές επιτροπές, τα λεγόμενα ΡΑΚ, για όλα τα θέματα που αφορούν την αλληλεία είναι σημαντικό και της διαχείρισης της αλληλείας. Πρέπει λοιπόν να αναγνωριστούν αυτές οι οργανώσεις, να θεωρηθούν ε, σημαντικός εταίρος και να έχουν φωνή. Ίσο ρόλο με τις άλλες οργανώσεις. Τέλος. δεν ξέρω αν και η συνάδελφος Άννα θα το παρουσιάσει. Α, το τελευταίο τότε αυτό για την ε, Γαλλικία θα το αφήσω για τη συνάδελφό μου. Παρακαλώ. Λίγη ησυχία παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που δόθηκε αυτή η σημασία στα θέματα φίλου. Έγραψα μια γνωμοδότηση για την Ρέτζι, για την αλληλεία μικρής κλίμακας και την παραδοσιακή. Το μελετήσαμε ως ομάδα σε βάθος. Το θέμα της συμμετοχής και της εργασίας των γυναικών στην αλληλεία είναι πολύ σημαντικό σε συγκεκριμένες αλληλευτικές ζώνες που οικονομικά εξαρτώνται πολύ από την αλληλεία σε πολλές περιπτώσεις είναι η μόνη δυνατότητα που έχουν πολλές γυναίκες για να εργαστούν. είτε ως ε, αποκλειστική απασχόληση ή ως ένα συμπλήρωμα για τις οικογένειές τους. Αλλά, όπως είπε και η κυρία Μπάουερ, δεν αντιμετωπίζεται από νομική άποψη, δεν αναγνωρίζεται όπως πρέπει. Ορισμένες φορές αναγνωρίζεται μερικά, οπότε παίζει ρόλο και για το επίπεδο της σύνταξης. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, τώρα στη Γαλλικία. Η παράκτια παραδοσιακή αλληλεία έχει να κάνει και με τις ε, υδατοκαλλιέργειες. Θα έπρεπε να γίνει αυτή η αναφορά στην εντατική υδατοκαλλιέργεια, γιατί οι γυναίκες που εργάζονται στην αλληλεία εργάζονται επίσης και στην οστρακοκαλλιέργεια. Δηλαδή τη συλλογή θαλασσινών. Αυτό γίνεται κυρίως από γυναίκες στη Καντάβρια, τη Γαλλικία και τη Βρετάνη. Επίσης οι γυναίκες επισκευάζουν τα δίχτυα στα λιμάνια. Δεν υπάρχει επαρκής επαγγελματική αναγνώριση. Σε πολλές περιπτώσεις η εργασία τους στη συλλογή οστράκων ή στην αλληλεία δεν πάσχει μόνο από αυτή την έλλειψη κοινωνικής αναγνώρισης και κοινωνικού περίγυρου, αλλά και από μόλυνση, από την έλλειψη υποδομών, από τις κλιματικές αλλαγές, από την αναγκαστική έλλειψη απασχόλησης, θέματα δημόσιας υγείας, τοξίνες για παράδειγμα, τοξικές ουσίες, τα απορρίμματα, ε, η μόλυνση από το πρεστίζιο από το έρικα, με πετρελαιοειδή κτλ. Οι γυναίκες στην Αλία χρειάζονται αξιοπρεπείς συνθήκες, επαρκές εισόδημα, αναγνώριση, επαγγελματική, σταθερότητα στην εργασία και πάνω απ' όλα χρειάζονται αναγνώριση ορισμένων ασθενειών γιατί θίγονται πολύ από ασθένειες ε, ρευματολογικές. Δεν αναγνωρίζεται αυτό ως επαγγελματική ασθένεια. Να το βάλει λοιπόν η συγκήτρια. Και τελευταίο. Υπάρχουν γυναικείς οργανώσεις όπως ε, η ΑΚΤΕΑ που είναι οι γυναίκες για την αλληλεία στην Ευρώπη που εργάζονται ενεργά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μια ένωση που έχει γίνει από γυναίκες που εργάζονται στην Αλία, από διάφορες χώρες, περιφέρειες κτλ. Η Επιτροπή που είναι εδώ παρούσα λοιπόν θα πρέπει να τη συμπεριλάβει στην νομοθετική διαδικασία και για το μελλοντικό Ταμείο Αλίες και το Θαλάσσιο Ταμείο για να μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται για θέματα πολιτικής ισότητας φύλων. Οι γυναίκες λοιπόν αυτές, πολλές, εργάζονται δωρεάν όλη τους τη ζωή ή με ελάχιστες συνθήκες ασφάλειας και υγείας και υγιεινής. Είναι ώρα επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει πόσο αξιοπρεπές είναι το επάγγελμά τους όπως οποιοδήποτε άλλο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Όχι άλλες παρεμβάσεις, δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις από τους συναδέλφους. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 29 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα. Η Επιτροπή μας θα ψηφίσει στις 24 Απριλίου και η Επιτροπή Αλία στις 30 Μαΐου. Ολοκληρώσαμε με το σημείο αυτό και με την ίδια την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και θα διακόψουμε για ένα λεπτό μέχρι να αρχίσουμε την επόμενη φάση της συνεδρίας.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 We will start now. Να ξεκινήσουμε τώρα. Καλώς ήρθατε όλοι. Does everybody hear me? Με ακούτε? You don't know? <laughs> okay, but it's, it's, it's a red sign. <laughs> Eh, I will swap. Είναι αναμένο το μικρόφωνο. Θα περάσω λοιπόν στα σουηδικά. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, φορέστε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Okay. Ναι, Καλωσορίζω θερμά όλους τους παραβρισκόμενους στη σημερινή συνεδρίαση με μεγάλη ε, χαρά μου θα ψηφίσουμε σήμερα για την τόσο σημαντική αυτή έκθεση. Χαίρομαι που βρίσκονται εδώ και οι συνάδελφοι της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, είναι εδώ και ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Θα του δώσω το λόγο πολύ γρήγορα για να μας ε, κάνει κάποια σύντομα σχόλια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Γκούσταυσον. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι πάλι εδώ. Είναι μεγάλη μου χαρά να συμπροεδρεύω ξανά μαζί σας. Η διαδικασία αυτή επικοδοματική συνεργασία μεταξύ των επιτροπών ε, στο σώμα μας, της Επιτροπής ΦΑΜ και ΛΥΜΠΕ, μας οδηγεί στο να προεδρεύουμε σε μια ψηφοφορία μαζί. Παρακαλώ, ε, προσέξτε να, αν θέλετε. Θα ασχοληθούμε με την ψηφοφορία και το μόνο που έχω να πω είναι ότι πάντοτε αυτέ του είδους οι διαδικασίες είναι επικοδομητικές. Τώρα ασχολούμαστε με την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, όπως παλιότερα είχαμε κάνει με την εμπορία ανθρώπων και με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας. Ευχαριστούμε λοιπόν εδώ τους εισηγητές, τις εισηγήτριες, τους σκιώδεις εισηγητές και εισηγήτριες για όλες τις προσπάθειες που έκαναν για να καταλήξουν σε συμβαστικές λύσεις. Ελπίζω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα μέσα από τη σημερινή ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μπορείτε να μιλήσετε όσο θέλετε και όση ώρα θέλετε, αλλά όχι μέσα σε αυτή τη συνεδρίαση. Εκτό αίθουσα, παρακαλώ. Ή τουλάχιστον κάντε λίγο ησυχία. Είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθεί κανεί στον ομιλητή. Να δώσω το λόγο στου ε, εισηγητέ. Δεν ξέρω ποιο θέλει να ξεκινήσει. Eh. Δεν θα μακρηγορήσω, διότι θέλετε να ψηφίσετε ώστε να τον πιο σύντομα η οποία είναι μακροσκελής, εργαστήκαμε σκληρά, πολύ καλή συνεργασία όπως είπε και ο Πρόεδρος η κυρία Παρνάλοβα και εγώ. Ευχαριστώ πολύ την γραμματεία, διότι πήραμε 500 τροπολογίες και καταλήξαμε σε βασικές τροπολογίες. Νομίζω ότι όλοι είχαν δυνατότητα να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στα θύματα αυτό που επιδιώκουμε. Δηλαδή να υπάρχουν ε, ελάχιστες προδιαγραφές στην Ευρώπη. Είναι μια σημαντική στιγμή. Τίποτα άλλο, κυρίως πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τα θύματα. Η κυρία Παρμάνοδα. Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ την κυρία Χιμένεθ, τους Κιώδης, τη Γραμματεία για την καρποφόρα συνεργασία. Ήταν δυσχερές το έργο μας να καταλήξουμε στους καλύτερους συμβασμούς. Ε, είχαμε 550 τροπολογίες, ούτως ώστε να συμπεριλάβουμε μια έκθεση που να έχει μια εσωτερική λογική. Ό,τι μπορούσαμε να συνδυάσουμε, το συνδυάσαμε Ό,τι μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε το συμπεριλάβαμε. Ένα σύντομο σχόλιο. Λόγω τεχνικών ζητημάτων μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να θεωρούν ότι δεν υποστηρίχθηκαν οι τροπολογίες τους. Αυτό σημαίνει γιατί καλύπτονται σε κάποιο άλλο σημείο με άλλο τρόπο. Όχι γιατί δεν εξετάσαμε την πρόθεσή τους ή ότι δεν θέλουμε να συμπεριληφθεί η άποψή τους. Είναι τεχνικό, όχι πολιτικό θέμα. Είμαι απογοητευμένη ιδιαίτερα που ορισμένες φορές ε, έτσι λειτουργεί η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους εργάστηκαν και ελπίζω η έκθεσή μας να είναι ιδιαίτερα δυναμική τελικά. Πρόεδρος, Πριν ξεκινήσουμε και περάσουμε στην ψηφοφορία, άλλοι δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο για διαδικαστικό. Να πω απλώ ότι θα πρέπει να είσαστε πολύ σύντομοι. Η κυρία Σαρχεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι συνοπτική. Εάν εμεί μπορούσαμε να επιλέξουμε ω πράσινοι, δεν θα γινόταν τώρα ψηφοφορία. Όπω είπε η συγγήτρια, ήταν τεράστιο το έργο μα, πάνω από 500 τροπολογίε που εξετάσαμε και μόλις πριν από μισή ώρα ολοκληρώσαμε τον κατάλογο της ψηφοφορίας. Το απόγευμα σήμερα χρειάζεται και να συμπεριλάβουμε πάλι κάποιες τροπολογίες που είχαν βγει από τον κατάλογο, διότι κάποιες άλλες θα μπορούσαν να εκπίπτουν. Δεν έχουμε αφιερώσει αρκετό χρόνο για να δούμε με προσοχή αυτό το νομοθέτημα και να ψηφίσουμε τόσο γρήγορα κάποιες συμβαστικές τροπολογίες αναγκαστήκαμε να τις βρούμε. Είναι, κάποιες άλλες 10-15 δεν βασίζονται σε καμία συμβαστική τροπολογία. Εδώ θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το αποτέλεσμα ως τριμερή βάση για τον τριμερή διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Οι πράσινοι θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετή η δουλειά που έχει γίνει. Θα έπρεπε να έχουμε κι άλλο χρόνο και να υπάρξουν συμβαστικές τροπολογίες για όλα τα σημαντικά άρθρα. Αυτό δεν ισχύει. Καταλαβαίνω ότι η ψηφοφορία θα γίνει ούτω ή άλλω, αλλά θέλουμε να σημειωθεί. Αυτό το νομοθέτημα, αυτή την νομοθετική πρόταση δεν την έχουμε πάρει αρκετά σοβαρά. Πιεζόμαστε για να πάμε στην ψηφοφορία. Eh, Ευχαριστούμε. Άλλοι δύο ε, συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Λόπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήμουν συνεισηγήτρια για το ένταλμα Ευρωπαϊκής Προστασίας για τις γυναίκες που είναι θύμα βίας. Παρουσίασα πολλές τροπολογίες και θα ήθελα να εξηγήσω. Ευχαριστώ για όλες τις τροπολογίες που συμπεριλήφθηκαν στις συμβαστικές, αλλά τονίζω ότι όλες οι δικές μου που δεν έγιναν δεκτές αφορούν τις γυναίκες που είναι θύματα κακομεταχείρισης στις χώρες όπου η κακομεταχείριση δεν θεωρείται ούτε καν αδίκημα. Όχι έγκλημα να θεωρείται. Οι γυναίκες αυτές είναι θύματα κακομεταχείριση. και αν εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται οι πράξεις αυτές από το αστικό δίκαιο, δεν θα μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε. Έγινε μεγάλη συζήτηση κατά τη διάρκεια της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Προστασίας αλλά δεν καταφέραμε να επιτύχουμε τίποτα για αυτές. Τονίζω λοιπόν ότι όλο αυτό το πακέτο βοήθειας για τα θύματα στην ουσία μπορεί να βοηθήσει μόνο τα, μέλη της οικογένειας των θυμάτων. Γιατί τα θύματα θα έχουν ήδη θανατωθεί. Μια, ορισμένες λοιπόν γυναίκες σε αυτές τις χώρες όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να διωχθούν ποινικά δεν θα μπορέσουν να βοηθηθούν από αυτό το πακέτο. Ευχαριστώ. Δεν ήταν ακριβώ διαδικαστικό, λέει ο πρόεδρο. Ε, αλλά θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Χιμένεθ για διαδικαστικό. Θα ήθελα να καθησυχάσω και να σας πω όλους και στην κυρία Παρμάνοβα με την οποία συνεργάστηκα ότι αυτή η έκθεση θα βοηθήσει όλα τα θύματα. Θα προσπαθήσει να τα βοηθήσει όλα τα θύματα. Είναι αδύνατο ή σχεδόν αδύνατο σε μία έκθεση για τις ελάχιστες προδιαγραφές να τους ευχαριστήσουμε όλους γιατί καταλαβαίνω ότι θεωρούν όλοι ότι είναι ευκαιρία αυτή η έκθεση αλλά εξηγήσαμε δεν είναι δυνατόν και δεν επιτρέπω και θέλω να απαντήσω στην κυρία Σαρχεντίνη δεν επιτρέπω δεν επιτρέπω κυρία Σαρχεντίνη να λέγεται ότι δεν αντιμετωπίσαμε σοβαρά το νομοθέτημα ή τα θύματα. Και κυρία Βεχερίλ, όλη μου τη ζωή την έχω αφιερώσει στο να υπερασπίζουμε τα θύματα. Δεν επιτρέπω να μου λέτε τέτοια πράγματα. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα βοηθήσουμε τα περισσότερα θύματα, θα το επιχειρήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να εργαζόμαστε υπέρ των θυμάτων. Δεν συμφωνώ λοιπόν με την κυρία Ρομέρο και την κυρία Σαρχαντίνη. Δεν μπορούμε όλα να τα αριθμίσουμε τώρα και με αυτό το νομοθέτημα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, αλλά μπορείτε να έχετε ίσχυ τη συνείδησή σα και να ψηφίσετε για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε. Και άλλο διαδικαστικό από τον κύριο Κροτσέτα. Μια, μια σύντομη διευκρίνηση. Επειδή οι συγητές αναφέρθηκαν στην προσπάθεια διαμεσολάβηση στο να βρεθούν συμβαστικέ τροπολογίε, πρέπει να πω ότι βρεθήκαμε στην άβολη θέση να είμαστε σκιώδει συζητητέ, δηλαδή να είμαι σκιώδη συζητητέ για την ομάδα μα και τελικά λάβαμε κάποιε προτάσει για να καταλήξουμε σε συμβαστική πρόταση. Νομίζω ότι αυτά τα βρίσκω πολύ σοβαρά όταν μιλάμε για προστασία θυμάτων. Εγώ θα ψηφίσω ανεξαρτήτως από τέτοιου είδους ε, σκέψεις και εκτιμήσεις. Ανεξάρτητες από αυτές που εξέφρασαν οι συγητές ή οι πολιτικές ομάδες. Για περιπτώσεις συλλογικών εκκληματικών πράξεων, θύματα τρομοκρατίας ή της μαφίας. Δεν έγιναν προσπάθειες για συμβαστικές τροπολογίες. Και τροπολογίες που έβαλα όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι βουλευτές. Ε, η διαφορά των φίλων είναι κάτι που έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Αν κάποιος πετάξει μια βόμβα, ας πούμε, σε έναν ε, δικαστή, το μόνο θέμα δεν είναι το φίλο, Πρόεδρος, θα έπρεπε να συντομεύεται. Ε, και πρέπει να προχωρήσουμε και με την όλη διαδικασία. Καταλαβαίνω ότι ήταν δυσχερέστατο το έργο σα, ήταν πάρα πολλέ οι τροπολογίε που υποβλήθηκαν. Οι προθεσμίε δεν επέτρεψαν να υπάρξει πολλή χρόνο, αλλά έχουμε το σχέδιο του καταλόγου ψηφοφορία. Δεν υπήρξαν σχόλια. Ε, την είδαν όλοι, πάλι δεν υπήρξε σχολιασμός. Υπάρχουν ισχύοντε κανόνε. Δεν βρίσκω να υπάρχει κάτι εξωσημείωτο στην όλη διαδικασία. Πιστεύω ότι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ θέλουν να γίνει η ψηφοφορία αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν ε, θα πρέπει να συμπεράνω. Οπότε, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, θα μιλήσω αγγλικά. Προ, προηγουμένως όμως, θέλω να πω ότι θα ήθελα το τεύχος αυτό του κατάλογου ψηφοφοριών να το δούμε με έναν τρόπο ιδιαίτερα προσεκτικό και να είμαι απολύτω δίκαιο. Αν γίνει κάποιο λάθο, αν κάτι παραλείψω, ε, παραλείψτε και εσεί να μου το επισημάνετε. Όλε οι προτάσει όπου υπάρχουν ε, αποκλίνουσε απόψει των εισηγητών θα ψηφιστούν ηλεκτρονικώ, κατευθείαν. Οπότε μην ζητήσετε έλεγχο, θα γίνει αυτομάτω. Οπότε, ας περάσουμε στην ψηφοφορία αυτή καθεαυτή. Θα μιλήσω αγγλικά για να διευκολύνω όλους σας. Να ψηφίσουμε τη συμβαστική πρόταση 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 2.14 εκπίπτει. Ψηφίζουμε την 2.12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, οι 213 και 21 εκπίπτουν. 215. Άρχεται η ψηφοφορία. And the, vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεν λειτουργεί το δικό μου το μηχάνημα. Μάλιστα. Τρία μηχανήματα δεν λειτουργούν, βλέπω. Ούτε το δικό σας. Τέσσερα. Ο τεχνικός θα μπορούσε να το κοιτάξει. We, we, we, do that again. Να ξαναψηφίσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικώς για την 215. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Όχι ακόμα. πέρα Εγκρίνεται. ...217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 218 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 220. Ε, εντάξει, ψηφίζουμε ηλεκτρονικώς για τη 219. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 220 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 221 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 222 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 226 ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 225. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 224. 224. Υπέρ. Όχι, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικος Άρχεται η ψηφοφορία για το 224. The vote is open and the vote is missing one. The vote is closed. Πέρας, εάν δεν προλάβατε. Εγκρίνεται. 228 υπέρ, κατά, αποχές, μάλλον πρέπει να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικός λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρα 221 και 230 εκπίπτουν. 227 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται απορρίπτεται 232 υπέρ 232 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 234 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 233. Όχι λάθος. 235. Ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 236 και 37 είναι πανομοιότυπες τροπολογίες, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 238 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 239 εκπαιδευτεί. 240 υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 241 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 242 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Συμβιβαστική πρόταση 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα, Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στη 243. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 251 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 254 δεν θα ψηφιστεί. 256. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 257. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς για τη 257. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is closed. Πέρασε. Εγκρίνεται. Σαφής διαφορά. 258 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 260 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 261 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 262 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δύο 264 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίθηκε. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. 264. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 265 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 267 υπέρ κατά εγκρίνεται 268 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική πρόταση 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Πιο κάτω. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 271, 272 και 273 εκπίπτουν. Όχι. Η 273 μένει. Ψηφίζουμε. 273 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς για τα 273. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Απορρίφθηκε. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 275 υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. 274 υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 276 υπέρ. Όχι, είναι πανομοιότυπε. Δεν χρειάζεται.

Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Άρα περνάμε στην συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 291. 291 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικός 291 υπέρ. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Απορρίφθηκε. Δεν χρειάζεται να σηκώνετε τα χέρια σας. Ή μάλλον όταν τα σηκώνετε να φαίνεται. 292 ε, εκπίπτει. 293 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 294 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. κατα αποχε εγκρινεται 294 ηλεκτρονικη ψηφοφορια αρχεται η ψηφοφορια περας Εγκρίνεται. 295 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 296 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμ... Τροπολογία 302. Ναι. 302. 302 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 303 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 304 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 305, όχι δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 308 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Καλά, θα το ελέγξουμε. 48 ηλεκτρονική ψηφοφορία και θα δούμε πώς να αλλάξω γυαλιά. Οπωσδήποτε θα πρέπει να αλλάξω. Έχω κάτι προβλήματα όραση, την είχα την υποψία, τώρα βεβαιώθηκα. 49. Σα ευχαριστώ όμω που είσαστε τόσο ε, δραστήριοι, τόσο ενεργοί. 49 υπέρ. Κατά. Τριακόσια «310 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 311 Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 309 επιπτή. 312 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε για την 312. 312 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, απορρίφθηκε. 313 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 318. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 319. Ας ελέγξουμε για 318. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. και δεν φορούσα καν τα γυαλιά μου, αλλά δεν ήταν σαφές. 319, υπέρ. Κατά, αποχές. Σαφώς απορρίπτεται. 53, υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Άρα, η 320 εκπληκτή 321, 321 υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 322. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3.25 εκπίπτει. Συμμεβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμμεβαστική 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. 329. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. 329. Πέρας. Εγκρίνεται. 332. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 333. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Σαφώ εγκρίνεται. 334. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 335. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. 335 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 336 ηλεκτρονικού και ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 337 υπέρ. Κατά. απόχέ. Νομίζω πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς για την 337. Έλεγχο λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρα η 341 εκπίπτει. 338 3.38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 339 339 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε 340 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος Έχω πάλι έκανα λάθος 340 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 342. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω και εδώ πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. 342. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν ανάπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 343. Εκπίπτει. 344 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 345 υπέρ, κατά, αποχές, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Όχι ακόμα. Όμω πέρασε παρόλα αυτά. Απορρίπτεται. 346 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 347 και 348 που είναι πανομοιότυπες. Από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 353 και 355 ε, είναι πανομοιότυπες. Από κοινού, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. 353-355. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με διαφορά. 354 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 356 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 357 ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. 350... 359, 359, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρα ψηφίζουμε την 360. 360 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 358 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 361 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 362 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 364 υπέρ. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 363 εκπίπτει. 365 και 367 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται μάλλον. 366. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 368. Υπέρ. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία μάλλον. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 369. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 370 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 371 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. It's, and the vote is closed. It's adopted. Πέρας. Εγκρίνεται. 374 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Άρα ψηφίζουμε για την 372. 372 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 377 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς για την 377. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 375 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 373. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πρέπει να ελέγξουμε. 373. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Άρα ψηφίζουμε την 376 Σωστά. Ναι. 376. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 378 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 379 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 380 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 381 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 382. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. 382. Πέρας. Εγκρίνεται. 383 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 384. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 385. Εγκρίνεται. Η 385 δεν θα ψηφιστεί. 386. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 387. 387 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 388 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 389. Είναι επανομοιότυπες. Με συγχωρείτε. 390. 390 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 391 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 392 ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 393 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 62. Πέρα. Εγκρίνεται. 394 δεν θα ψηφιστεί. 395 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 396 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 397 Υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικό για την 63. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται δεν σηκώνεται αρκετά ψηλά τα χέρια. 16. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 403. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. now we have an oral amendment. Προφορική τροπολογία τώρα. Να ρωτήσω, έχει κανείς αντίρρηση. Να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Όχι. Ωραία. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Ηλεκτρονικά. 405. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η, 4, η 404 καταπίπτει. Πάμε στην 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν κατάλαβα καθόλου. Πάλι. Ποιος είναι υπέρ. 65. Κατά. Αποχές. Ε, γκρίνεται προφανώς. 406. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 407. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 408. Όχι. 409. 409. Η 408 δεν θα ψηφιστεί. 409 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε να ψηφίσουμε την 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Πάμε στην 410. 410. Θα ψηφίσουμε την 410. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 411. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 412. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 413. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε την 413 λοιπόν ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 414. Άρχεται η ψηφοφορία για την 414. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε και εδώ. 414. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 415 αποσύρεται, 416, 416 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 68 υπέρ, κατά, αποχές. 417 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 418. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 418. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 69, η 419 και η 420 είναι Όλε όλες μαζί λοιπόν. Υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνονται. Οι 70 και οι 422 ψηφίζονται από κοινού. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα εγώ. Λοιπόν, 70 και 422. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η 421 καταπίπτει. Πάμε στην 424. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την τροπολογία 71. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 425. Καταπίπτει. Πάμε στην 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 426 καταπίπτει. Πάμε στην 427. Ψηφίζουμε 427. Υπέρ. Κατά. Α, συγγνώμη, ναι, ηλεκτρονικά πρέπει να την ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε την 427 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 428. Επίσης ηλεκτρονικά. Υπέρ. Ε, ψηφίζουμε, συγγνώμη. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 429. Επίσης ηλεκτρονικά. Αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 430. Ηλεκτρονικά. Αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 432. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. «Ψηφίζατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 431. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 433. Υπέρ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, ηλεκτρονικά πρέπει να την ψηφίσουμε. 433 λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 435. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, να το ελέγξουμε, να το ελέγξουμε, συγγνώμη. 435 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 438 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 439 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 440 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 441. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 442 καταπίπτει. Ψηφίζουμε την 444. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 445 καταπίπτει, 446, 446 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 447 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 436 καταπίπτει, πάμε στη συμβαστική 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 442. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στην 453. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 455 καταπίπτει. Άρα 456 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η 76 καταπίπτει. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 457 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Την 457. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 19. Α, συγγνώμη. 462. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα πάμε στη συμβαστική 19. Προφορική τροπολογία. Έχει κάποιος αντίρρηση? Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν τη συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 463. Επίσης προφορική τροπολογία. Έχει κάνει αντίρρηση. Όχι. Ψηφίζουμε την 463. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 464. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 465. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 81 έχει αποσυρθεί. 466. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε μόνο το κείμενο που αφορά την προσθήκη στην τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν την 466. Μόνο αυτό το κείμενο της προσθήκης. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 467. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 467. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 469 καταπίπτει. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 470. Άρχεται η ψηφοφορία για την 470. Πέρας. Εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84. Υπέρ. 84 πάλι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 471. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85. Υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 472 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 473 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 474 ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 474. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 475. Πάλι ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 480. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 480. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 87. Ηλεκτρονικά. Στο δικό μου χαρτί έχει συν πλην. Εν πάση περιπτώσει, ε, ε, ό,τι και να έχει, δεν Πάμε στην 481. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 482. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 484. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 485. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 486. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 486. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 88 καταπίπτει. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 487. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για 487. Πέρας. Εγκρίνεται. 488. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 488, 68, συγγνώμη, καταπίπτει. 489. Υπέρ. Εγώ έχω άλλο κατάλογο. Δεν λέει στο δικό μου το κατάλογο ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εν πάση περιπτώσει, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 489. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 4.90. Επίσης ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 4.91. Επίσης ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 483 καταπίπτει. Πάμε στην 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 492. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 493. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 494 ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 494 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 495 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Α, συγγνώμη, είναι προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση. Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν την 495. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 496 δεν την ψηφίζουμε. 497 ψηφίζουμε τη 497. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 498 λοιπόν καταπίπτει. 500 ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 500 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 499 λοιπόν εκπίπτει. 501 ηλεκτρονικά. Πέρας. Ooh, it's adopted. Ε, compromise 20. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 505. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 506. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 506. 506. 506. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 510. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 512. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 513. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, να το ελέγξουμε. Μάλιστα. 513. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 514. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Την 514. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 515. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 516. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 518. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Check. Check on file. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 518. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is... It was closed. It's adopted. Πέρας. Εγκρίνεται. 520. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 520. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 521. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 525. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 526. Υπέρ. Α, συγγνώμη. Σε δύο μέρη. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της 526. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στο δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5.27 Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5.28 Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96 Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, εγκρίνεται, εγκρίνεται εννοούσα, εγκρίνεται εννοούσα, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εννοούσα εγκρίνεται. Λάθος. Γράψτε λάθος. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 529. Ε, Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 529. The vote Πέρας. Εγκρίνεται. Να κάνουμε ένα για καφέ τώρα. Και τι, κανένα μπισκοτάκι, κανένα βούτυμα, κάποιος κάτι. Λοιπόν, πάμε στην 530. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90... 98, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 531 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 532 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 533 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην τροπολογία 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103. Υπέρ. Α, συγγνώμη. Ούτε αυτό το λέει όμως ο καταλογός μου. Μάλλον έχω λάθος κατάλογο. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την τροπολογία 103. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν την 104. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Στο δικό μου το κατάλογο λέει ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 105. Ωραία. Ηλεκτρονικά λοιπόν ψηφίζουμε την 105. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 107. 107. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Την 115. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 120 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 121. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 122. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 130. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 130. And the vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 8 και την 131 από κοινού, διότι είναι ταυτόσημες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές, συμβιβαστική 29 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Πάμε στην 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 138. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, να το ελέγξουμε. Μάλιστα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 138. Άρχεται η ψηφοφορία. It's rejected. Απορρίπτεται. Η 139 εκπίπτει. Όχι. Ψηφίζουμε την 139. Ψηφίζουμε την 139. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 141. Υπέρ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν την ψηφίζουμε την 141. Συμβιβαστική 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 146. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 146. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 149. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 149. Πέρας. Εγκρίνεται. 151. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 152 ηλεκτρονικά. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 156. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 160. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 160. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 33. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Πάμε στην 164. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 164. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 165. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 34. Είναι προφορική τροπολογία. Έχει κανείς αντίρρηση? Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν την 134. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 168. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Από ό,τι μου φάνηκε σαν να απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Εγκρίνεται. 169. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία σε τμήματα για την 170. Να τη δούμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Άρχιδη ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της 170. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα εκπίπτει. Και το τρίτο εκπίπτει. Πάμε στη 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρα η 18 καταπίπτει και η 171 επίσης πάμε στη 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εγκρίνεται συγγνώμη η 173 καταπίπτει πάμε στη συμβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην 181. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 182. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. βασική 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Yeah. And then we have electronic vote on 108. Πάμε στην 187. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 187. And the vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβιβαστική 37. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 190. 190. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Η το 191 δεν την ψηφίζουμε. Πάμε στην 192. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 193 in favor. 193 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 22 καταπίπτει. Πάμε στην 23 υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε μάλλον. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 23. The Πέρας. Πολύ περίεργο αποτέλεσμα. Εγκρίνεται, με πάση περιπτώσει. Πάμε στη συμβαστική 38. 38. Η 194 είναι ταυτόσιμη με την 23. Α, συγγνώμη. Λάθος μου, λάθος μου. Δεν το είπα. Πάμε στη συμβαστική 38 λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 197. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 201. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 202. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 203. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 204. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 205. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 206. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εντάξει, ας την, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω όμως ότι εγκρίνεται. Σηκώνετε τα χέρια σας καλά, παρακαλώ. Εγκρίνεται λοιπόν. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται ε, τροπολογία 207 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται περνάμε στην γνωμοδότηση της ε, νομικής τζούρι Yeah. to... Λοιπόν, θα τις ε, ψηφίσουμε όλες μαζί μέχρι τη 17. Εντάξει. Κυρία Γιάννα Εντάξει. Α, καταπίπτουν. Δεν έχουμε να ψηφίσουμε η 15 είναι η πρώτη την οποία πρέπει να ψηφίσουμε. Όλες οι άλλες έχουν ήδη καταπέσει. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 όλες καταπίπτουν. Περνάμε λοιπόν στη 15. Α, όχι, συγγνώμη, και την 11. Πρέπει να την ψηφίσουμε γιατί είναι προσθήκη. Ψηφίζουμε την τροπολογία 11. 7 έως 10 καταπίπτουν. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Οι τροπολογίες 12 και 13-14 καταπίπτουν. Ψηφίζουμε τη 15. Υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 16 καταπίπτει. Ψηφίζουμε τη 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται. Η 19 Ωραία, με συγχωρείτε. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 18. Άρχεται η ψηφοφορία. 18. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 20. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε την 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ πάλι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 22, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 23, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 25. Α, ναι, 25. 25, υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται δεν θα ψηφίσουμε δεν χρειάζεται να ψηφιστεί 24 25 ψηφίζουμε εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 έως 32 καταπίπτουν. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία, να ελέγξουμε 35. Άρχεται η ψηφοφορία για την 35. Απορρίπτεται. πίπτη 36. Τροπολογία 36 υπέρ. 37 συγγνώμη. Υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 39. Άρχεται για την 39. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Σαράντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 καταπίπτει. δύο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σαράντα τρία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σαράντα τέσσερα, υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται. Ελέγχουμε τη 44, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 45 καταπίπτει, τροπολογία 1, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3 καταπίπτει, τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Ωραία, να κάνουμε έλεγχο για την 4. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 4. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 νομίζω καταπίπτει η τελευταία. Η τελευταία. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Σαφώς εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος, άρχεται η ψηφοφορία για το σύνολο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται, σαφώς. Συγχαίρω τους εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ.